κινηματογράφου στην ψηφιακή εποχή. Τέσσερα λεπτά έχει το λόγο ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε επίτροπε, στη σημερινή μου παρέμβαση θα κυριαρχήσει ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Ε, τα τελευταία χρόνια είδαμε μεγάλη επιτυχία του ευρωπαϊκού κινηματογραφικού χώρου. Είχαμε παραγωγή πάνω από χίλιων ε, ταινιών, αλλά ο αριθμός ε, των θεατών που είδαν τις ευρωπαϊκές ταινίες είναι αντιστρόφως ανάλογος των ταινιών που παράγονται. Κατά κύριο λόγο, οι ταινίε προβάλλονται στη χώρα στην οποία παράγονται. Πολύ συχνά δεν βρίσκουν κοινό αυτές οι ταινίε και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προωθήσουμε την, ε, ε, τις ταινίε, διότι είναι ένας τρόπος να υπάρχει πολιτιστική ποικιλομορφία και να μάθουμε τους γείτονές μας. Γι' αυτό ακριβώς η έκθεσή μου για την διανομή των ευρωπαϊκών ταινιών είναι πάρα πολύ σημαντική. Πέραν των ε, κινηματογραφικών αιθισών που είναι ο χώρος που επιλέγει κάποιος για να δει μια ταινία, υπάρχουν και άλλοι τρόποι διανομής μια ταινία χάρη στην ε, ψηφιακή εποχή. Υπάρχει χώρος για καινοτομία εδώ και για μεγαλύτερη ελαστικότητα. Ο ευρωπαϊκός ε, κλάδος του κινηματογράφου θα πρέπει να αναζητήσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέα διάβλους διανομής εκμεταλλευόμενο και τις ε, διασυνοριακές υπηρεσίες και ε, εγγυόμενοι έτσι στους Ευρωπαίους ε, θεατές μεγαλύτερη επικοινομορφία χάρη στην δυνατότητα να υπάρχουν διαφορετικά μέσα διάδοσης των ταινιών. Χρειάζεται όμως να δημιουργήσουμε ευνοϊκό κλίμα ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τον κατάλληλο οικονομικό και πολιτισμικό ιδανικό χώρο που θα δημιουργήσει ε, κίνητρα για επενδύσει και να μπορέσουμε έτσι να θεμελιώσουμε την πολιτισμική ποικιλομορφία. Θα πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των ταινιών που ε, υποτιτλίζονται τώρα ε, στοιχίζει πολύ φθηνότερα ο υποτιτλισμός χάρη στην ε, ψηφιακή υποστήριξη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να προωθήσουμε καταλήλωση ταινία. Όπως επίσης σημαντικά είναι και τα διάφορα φεστιβάλ κινηματογράφου όπως το φεστιβάλ των Κανών του Βερολίνου χάρη σε αυτά μπορούμε να έχουμε ένα διευρωμένο ευρωπαϊκό κοινό η ταινία «Ίντα» του Παυλικόφσκι, την οποία είδαν λιγότεροι ε, θεατές στην Πολωνία, αλλά χάρη στη μεγάλη της επιτυχία είδαν πολύ περισσότεροι ε, οι Ευρωπαίοι ε, θεατές ε, και μετά από όλα τα βραβεία που έλαβε η ταινία το είδαν και οι Πολωνοί θεατές. Ε, αυτό μας δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Πρέπει όμως να υπάρχει και κατάλληλη χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα Media, το πρόγραμμα Connecting Europe θα μπορούσε να βοηθήσει, θα μπορούσε να υπάρχουν βέβαια και αλλά και από το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο ε, Χρηματοδότησης ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προώθησης, να υπάρχει διεθνής διανομή των ταινιών για να μπορέσουν να τις δουν όσο το δυνατόν περισσότεροι θεατές. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει και κατάλληλη εκπαίδευση του κοινού στο σινεμά. θα πρέπει να ξεκινούμε ε, από όλο και νεότερους μαθητές και σπουδαστές. Βεβαίως θα πρέπει να γνωρίζουμε σε ποιον θα ε, στοχεύσουμε, διότι πρέπει να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας ευρωπαϊκή ε, κληρονομιά κινηματογράφου. Θα πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα των κινηματογραφικών ταινιών για να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό αρχείο. Ε, η έκθεσή μου ε, αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή για να μπορέσουμε να έχουμε έναν ευρωπαϊκό πραγματικό κινηματογράφο και να υπάρχουν κατάλληλα μέτρα, διότι όλο ο οπτικοακουστικό τομέα περιμένει να δει και τι θα κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί του στήματο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Βέντα. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πρέπει να σταματήσουμε στις 11. Είπα ότι θα δώσω το λόγο σε κάποιους ακόμη. Ε, τώρα ε, έχω συναδέλφους, δύο που δεν έλαβαν το λόγο. Οι συνάδελφοι Καπούτο και Εντενόλφοι. Ο συνάδελφος Καπούτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η ενίσχυση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και ε, είναι ένας βασικός στόχος για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη ανάπτυξη της δυνατότητας της δημιουργίας. Αυτά εκφράζονται στο μέγιστο βαθμό στα κινηματογραφικά έργα όπου έχουμε ε, το συνδυασμό πολλών δεξιοτήτων. Εδώ σε αυτόν τον ορισμό θα πρέπει να προσθέσουμε και την ε, πολύ σημαντική οικονομική συνεισφορά. Ο τομέα οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασία και κυρίω σε μια ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη. Το καλλιτεχνικό λοιπόν σύστημα πρέπει να ε, ε, διαθέτει κατάλληλη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, ιδίω για δημιουργού μεγάλη εμβέλεια. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ανάπτυξη με τη χρήση τεχνολογιών ενό πραγματικού ψηφιακού ενεργειακού ρεαλισμού που θα μας βοηθήσει να έχουμε προστασία των ε, πνευματικών δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής. Κάποιες φορές το ένα, κάποιες φορές το ε, άλλο και κάποιες φορές και τα δύο. Θα πρέπει να υπάρχει προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και της ιδιωτικής δικαιωμάτων ζωής και θα πρέπει ίσως να συσταθεί και μια επιτροπή που θα ασχοληθεί με τον ορισμό του καλλιτεχνικού έργου το 2015. Ευχαριστώ κύριε Καπούτη, κυρία Ντενόλφη. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Από τις σπουδές Μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, από τις σπουδέ μου γνωρίζω πολύ καλύτερα τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν ε, κάποιοι στον οπτικοακουστικό τομέα. Για παράδειγμα, το να αναγνωριστούν ε, πολιτιστικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την άποψή μου, μέχρι τώρα δεν έχει ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα θέματα. Το κινηματογράφος και τα ευρωπαϊκά έργα ε, αντί να προστατεύσει το παραγωγικό μας σύστημα, επιτρέπουν παρεκκλώσεις ε, στην υποχρέωση να δίνονται το 10% των εσόδων ε, στην παραγωγή ευρωπαϊκών έργων. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, η αρχή που εγγυάται τις παραγωγές επέτρεψε παρέκκληση εκατομμυρίων ευρώ υπέρ, μιας, υπέρ της πολυεθνικής Walt Disney, η οποία ε, δεν επιτρέπει να βρουν ε, κατάλληλες ποιοτικές παραγωγές οι οποίες θα πρέπει να ε, μεταδίδονται στα κανάλια της. Αυτό είναι εις βάρος και στον εργαζομένο μας. Ο κινηματογράφος είναι κοινωνικό έργο καταρχάς. Και επομένως καθήκον μας είναι να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και να δημιουργήσουμε μια ενιαία ψηφιακή αγορά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Ο, κύριος, ε, ο Επίτροπος Χόγκαν. Ευχαριστώ. Ε, η Επιτροπή χαιρετίζει την υποστήριξη του Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βέντα, ο οποίος ετοίμασε αυτήν την έκθεση. Ο τομέας ο κινηματογραφικός είναι σημαντικός και οι προσανατολισμοί για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο είναι πάρα πολύ σημαντικοί το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή αναγνωρίζουν την αξία των ταινιών και ε, βεβαίως ε, ε, έχουμε ε, το 2013 1.346 ε, έργα παρήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ μικρό ποσοστό προβλήθηκε εκτός των χωρών παραγωγής. Βεβαίως αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες λόγω της ποικιλομορφίας πολιτιστικής και γλωσσικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ συχνά χρηματοδοτούνται από δημόσια κονδύλια και έτσι ε, δεν μπορούν να υποτιτλιστούν. Θα πρέπει ε, να αναπτύξουμε νέους ε, τομείς, να επωφεληθούμε την ψηφιακή τεχνολογία. Η Επιτροπή θα ήθελε διάλογο με την Ένωση η οποία θα ήθελε να καλύψει το χάσμα Υπάρχουν διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείε και διάφορες ομάδες σε πάρα πολλές τοποθεσίες ώστε να μπορέσουμε να δούμε την αποτελεσματικότητα, να υποστηρίξουμε τον τομέα, να αναπτύξουμε νέα business models λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή επανάσταση, να Ενθαρρύνουμε τον διάλογο με τον τομέα των οπτικοακουστικών ε, υπηρεσιών και να λάβουμε υπόψη την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και το φόρουμ επίσης ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε διασκέψεις, σεμινάρια, εργοτάξια ε, και τα πρώτα αποτελέσματα του φόρουμ θα λάβουν χώρα στις ε, Βρυξέλλες ε, το επόμενο έτος βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει σε αυτήν την διαδικασία ε, θα ήθελα επίσης να επισύρω την προσοχή σας πάνω στο πρόγραμμα Creative Europe Δημιουργική Ευρώπη που ασχολείται διασυνοριακά με τις ταινίε, με την διανομή, την προβολή με το δίκτυο Europa Cinemas και επίσης με, υποστηρίζεται επίσης ε, η υπηρεσία των VOD, των καταπαραγγελία βιντεοτενιών των υπηρεσιών βιντεοπαραγγελίας που δίνουν κίνητρα στον τομέα για καινοτομία ως προς την διανομή και διάθεση των έργων. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι ιδιώτες επενδυτές και να μην βασίζουν τόσο πολύ σε δημόσια κονδύλια. Όσο προς ε, τις ε, δημιουργικές ε, υπηρεσίες θα έχουμε αυτό το νέο χρηματοδοτικό μέσο για, στην αρχή του επομένου έτους. Κύριε Πρόεδρε, με την επανάσταση ψηφιακή θα πρέπει ο τομέας ο κινηματογραφικός να είναι στην πρωτοπορία της καινοτομίας. Η Δημιουργική Ευρώπη το πρόγραμμα θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία αυτή τα επόμενα έτη. Ευχαριστώ Επίτροπο και συζήτηση και αυτή